Περνάμε τώρα στο πρόγραμμα εργασία. Οριστική πρόταση του ημερησία διάταξη αποθετήθηκε στι 30 Ιανουαρίου διάσκεψη του Προέδρου. Ε, στι 19 Ιανουαρίου από τη διάσκεψη του Προέδρου. Θέλει κάποιο από αυτό το λόγο. Όχι. Θα ήθελα λοιπόν να σα προτείνω. Η συζήτηση για τα συμπεράσματα του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 30 Ιανουαρίου 2012 θα λάβει τώρα από τις 3 και 10 έως τις 5 παρα 20 χώρα. Η ώρα των ερωτήσεων προς την είπα το εκπρόσωπο θα γίνει 5 παρα 20 έως 6 παρα 20 και οι επόμενες συζητήσεις θα αρχίσουν στις 6 παρα 20. Η συζήτηση για την έκθεση του Οργαίζα Αγγουλό για την εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα θα αναβληθεί μέχρι την 5η. Η επιρώτηση για την προφορική ερώτηση για την εφαρμοσιμότητα της, ε, ε των, ε, των, των, των ομολόγων σταθερότητα θα ανεκατασταθεί από την Τουρκάζη Άγκολο. Επίσης θα έχουμε μια συνολική παρουσία της έκθεσης ΡΕΚΒΑ και η πρόταση ψηφίσματος για την ε, προσθέμενη αξία που προσθέτει ε, προτείνει το, η Επιτροπή Περιβάλλοντος σύμφωνα με το 88-2 θα περάσει αμέσως στην ψηφοφορία. Αν διαφωνεί κανένα. όχι βλέπω όλοι ενθουσιώδει, υπέρ, αποφασίζεται αυτό. Και τροποποιείται έτσι η μεσαία διάταξη. Περνάμε τώρα στις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της για